λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να κάνουμε μια δοκιμή. Δοκιμαστική ψηφοφορία δηλαδή. Οπότε βάλτε την κάρτα σας στο μηχάνημα, ε, αρχίζει η ψηφοφορία, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Δεν έχει κλείσει ακόμα η ψηφοφορία. Τι έγινε, έχουμε πάρα πολλούς που ψηφίζουνε. Και πείτε μας, για ποιο ψηφίζουμε. Α, δοκιμαστική Είσαστε κατά, οπότε εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν. Περνάμε στην κανονική ψηφοφορία, πρώτη ψηφοφορία. Ωραία, δεν είναι εδώ κορτιά, είπα εγώ. Λοιπόν, είμαστε στο σημείο 10, διορισμός Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. εγκρίνουμε τον ορισμό της κυρίας Κριστίν Λαγκάρτ ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά με μυστική ψηφοφορία. Οπότε, μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Τα νούμερα είναι εντάξει. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 37 υπέρ, 11 κατά, 4 αποχές. Συγχαρητήρια. Περνάμε στο επόμενο σημείο, σημείο 11. Πρόκειται για το διορισμό Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχει μια προφορική τροποποίηση όμως που προτείνεται. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας που για πρώτη φορά έχουμε μία γυναίκα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όμως είμαστε ακόμα πολύ μακριά από την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στους οικονομικούς, νομισματικούς και δημοσιονομικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι, οι γυναίκες αποτελούν την εξαίρεση, ιδιαίτερα στα υψηλά επίπεδα. Οπότε χάνουμε προσόντα, ικανότητες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό έχει δεσμευτεί υπέρ των γυναικών, χωρίς όμως συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και εμείς που έχουμε κληγεί πρόσφατα πρέπει να επιβεβαιώσουμε αυτήν την δέσμευση υπέρ των γυναικών σε υψηλές θέσεις. Υπάρχει και η Επιτροπή Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Λοιπόν, για το Εποπτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προτείνω μια τροπολογία από το Renew που λέει ότι ζητάει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εφαρμόσει την αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών στις διευθυντικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η τροπολογία αυτή πρέπει να σας πω δεν ε, έχει να κάνει με τον υποψήφιο. Είναι μια θεσμική αρχή όμως που θέλουμε να τηρείται. Και στα αγγλικά ε, η τροπολογία λέει τα εξής. Επαναλαμβάνω, η Μιλήτρια ζητάει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να βελτιώσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις ε, διάφορες ε, εκτελεστικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρακαλώ, Μάρκος. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι ε, θα προτιμούσαμε και θα μπορούσαμε να έχουμε πρόεδρο και του υποπτικού ε, οργανισμού αν είχε καταθέσει υποψηφίως κάποιος από τους φιλελεύθερους εφόσον το θέλανε τόσο πολύ. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία γυναίκα που να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Η κυρία Λάουτεν Σλίγκια μέχρι τώρα ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της πρότεινα να παραταθεί η και δεν ήθελε. Ως εκ τούτου ε, δεν είναι εύκολο να γίνει τίποτα. Και ε, το τρίτον, ε, θα ήθελα να πω στη συνάδελφο που διάβασε αυτό που διάβασε προηγουμένως, ότι σε ένα εδάφιο του ψηφίσματος αναφέρεται ήδη ότι θα πρέπει να υπάρχει ισότητα των δύο φύλων. Δεν ξέρω τώρα γιατί ε, θα πρέπει να το επαναλάβουμε. Αναφέρεται μία φορά και θέλουμε να το επαναλάβουμε. Και το τρίτο που θέλω να πω, ακόμα και αν είπατε ότι είναι προφορική τροπολογία, εδώ στο Κοινοβούλιο ήθιστε τέτοιου είδους ε, προτάσεις ε, να καταβάλλονται εκ των προτέρων σε γραπτή μορφή. Εγώ ήμουν συντονιστή, δεν πήρα τίποτα και είδα ότι αυτό που είπατε το είχατε στείλει μόνο στους συνεργάτες της πολιτικής ομάδας, άρα δηλαδή θα έπρεπε να είναι δυνατόν ε, πριν από την ψηφορία να έχει κανείς μπροστά του ε, προφορική τροπολογία για να ξέρει τι ψηφίζει. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους στο μέλλον να τηρούμε αυτούς τους κανόνες, γιατί ξέρετε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εργαστούμε εάν έρχεστε την τελευταία στιγμή, παρουσιάζετε μία προφορική τροπολογία και καλούμεθα εμείς να σκεφτούμε τι είναι ακριβώς αυτό. Καλύτερα να το έχουμε μπροστά μας σε γραπτή μορφή. Γι' αυτό εγώ είμαι κατά αυτής της προφορικής τροπολογίας. Υποθέτω ότι δεν πρέπει να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες. Αν θέλετε να πείτε κάτι, πολύ σύντομα παρακαλώ. Αλλιώ ας προχωρήσουμε στη διαδικασία και να αποφασίσουμε επί τη τροπολογία. Αλλά αφού μίλησε ο Μάρκο και εσεί έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Θέλω σύντομα να παρέμβω για να στηρίξω την τροπολογία αυτή και να αντιδράσω στην προηγούμενη παρέμβαση. Το να ακούμε ότι δεν υπάρχει γυναίκα για αυτή την θέση ε, δεν μου φαίνεται καθόλου καλή τοποθέτηση. Τόσες γυναίκες υπάρχουν εδώ πέρα, τόσες γυναίκες ασχολούνται με τα οικονομικά και με τα δημοσιονομικά. Δεν μπορεί να είναι αυτή η απάντηση. Στηρίζω λοιπόν την τροπολογία της συναδέρφου θα τη στηρίξουμε και ζητάω η Επιτροπή μας να είναι προσεκτική σε αυτά τα θέματα της ισότητας στο μέλλον, γιατί είναι πολύ σημαντικά και για τα δημοσιονομικά. Πρόεδρος, μην ξεκινήσουμε τώρα συζήτηση. Λοιπόν, ποιος είναι κατά της προφορικής αυτής τροπολογίας. Παρακαλώ να βλέπω χέρια, για να τάσω στις χειρός. Χρειαζόμαστε τέσσερις, είναι περισσότερο από τέσσερις αυτοί που αντιτίθεται. Οπότε δεν θα ψηφιστεί η τροπολογία αυτή. Και έτσι συνεχίζουμε και περνάμε στον ε, διορισμό του κύριου Μέρς στη θέση του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και πάλι η ψηφοφορία αυτή θα γίνει με μυστική ψηφοφορία. Και γρήγορα γιατί έχουμε και άλλες ψηφοφορίες. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη φοφορία. Α, από το ΕΛΚ είχαμε έναν παραπάνω που ψήφιζε. Τώρα είναι εντάξει, ωραία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 35 ψήφοι υπέρ, 14 κατά και 4 αποχές. Συνεχίζουμε και περνάμε στο τελευταίο σημείο, που είναι το σημείο 12. σχέδιο γνωμοδότηση Γενικός προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό έτος 2020 όλα τα τμήματα. Συμβαστική α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εδώ πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά και να σηκώνετε καλά τα χέρια αν θέλετε να πάμε πιο γρήγορα. Λοιπόν, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Και πάλι πρέπει να ελέγξουμε. Δεν ψηφίζετε; Ηλεκτρονικά λοιπόν θα ψηφίσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε και πάλι. Αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 15. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική γάμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Οι σοσιαλιστές είναι υπέρ. Ωραία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική δέλτα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνονται. Περνάμε στο δεύτερο κομμάτι. Που είναι τροπολογίες επί του προπολογισμού. Εδώ είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. Ξεκινάμε με την οίκον 6102 δεύτερη στήλη, έτσι. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. εγκρίνεται. 61.03. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61.04. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. εγκρίνεται. 61-22, Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61-37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61-20 υπέρ, κατά, αποχές, είναι υπέρ οι σοσιαλιστές, ωραία, εγκρίνεται. 61-00 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61-35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61-05 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61-06 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61-07 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61-08 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61-09 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61-10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61-24. Εδώ έχουμε μια προφορική ε, τροποποίηση. Φαντάζομαι ότι την έχετε, όχι. Σβέν, από ό,τι φαίνεται δεν έχει κυκλοφορήσει. Είναι μια γνωστή η τροπολογία με τη συνήθη διαδικασία. 61-24 λοιπόν στον κατάλογό μου όντω αναφέρεται η τροπολογία. Μα τη συζητήσαμε και στην ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στην Επιτροπή και συμφώνησαν όλες οι πολιτικές ομάδες που ήταν παρούσες. λέει αποθεματικό 1 εκατομμύριο αντί για 2 εκατομμύρια ευρώ όπως είχε κατατεθεί αρχικά. Θα ψηφίσουμε αν υπάρχει ένσταση. Υπάρχει καμιά αντίρρηση να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Η γραμματεία μου λέει ότι έχει μοιραστεί. πάση περιπτώσει, μοιράστηκε όπως έπρεπε να έχει μοιραστεί. Ποιος ξέρει, λοιπόν, υπάρχει καμιά αντίρρηση να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Όχι, λοιπόν, υπέρ της τροπολογίας με την προφορική τροπή. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 61-21. Υπέρ, κατά, αποχές. Εδώ θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 61-26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι σοσιαλιστές υπέρ. Εγκρίνεται. 61-27 υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 61-28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61-34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61.01 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61.36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61.11 και 61.17 που είναι ίδιες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 61.12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61.13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61-18 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, πέρα στις προφορίες. Εγκρίνεται. 61-29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61-14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61-15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61-16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61-30 με προφορική τροποποίηση πάλι, ίδια με την προηγούμενη. Ψηφίζουμε λοιπόν με την τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61-31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61-32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61-33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το τροποποιημένο κείμενο. Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Οι συντονιστές παρακαλώ για τρία λεπτά. Για ελάτε για να συμφωνήσουμε για την επόμενη συνεδρίαση. Κατά τα άλλα, σας ευχαριστώ πολύ για όλη την ημέρα που ήσασταν εδώ. Αύριο στις 9 θα συνεχίσουμε.